για την προστασία των ε, ζώων και την φυτογειονομική προστασία. Ε, Τρει μήνε έχει το Κοινοβούλιο για να εκφράσει άποψη για το θέμα αυτό που ξεκινάει από αύριο στι 20 Ιανουαρίου 2017.